για μια στρατηγική της ευζοίας των ζώων για το 2016-2020 και αυτό προέρχεται από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και χαιρετίζω τον κύριο Ανδρουκάητη στη συζήτηση και δίνω το λόγο στους συντάκτες αυτής της ερωτήσεως, τον κύριο Σικόρσκι από την Επιτροπή Γεωργίας για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να θέσω καταρχήν ένα ερώτημα προς την Κομισιόν που να συνάπτεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την ευζοία των ζώων μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2016-2020. Η ανακοίνωση της Κομισιόν για τη στρατηγική αυτή έχει τύχει θετικής απήχησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έχει θεσπίσει ένα, σαφές, ένα σαφή οδικό χάρτη για την προστασία της ευζοίας των ζώων. <clears throat> Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, τονίζει ιδιαίτερα τέσσερα σημεία στην, ε, στο ψήφισμά του του 2010 που έχουν μεταφερθεί στη στρατηγική της Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τις πρόοδους που έχουν <clears throat> επιτευχθεί μέχρι στιγμής και ζητά από την Κομισιόν σε σχέση με τους στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα να κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες. Το ερώτημά μου όμως είναι το εξή. Η Κομισιόν στο διάστημα 2016-2020 θα ακολουθήσει μια νέα στρατηγική για την προστασία και την ε, ευζοία των ζώων ώστε να μπορέσουν αυτά τα μέσα, αυτά τα μέτρα να ε, επιτευχθούν και να υπάρξει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι συνεκτική. Η στρατηγική προστασία των ζώων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι μια στρατηγική που περιλαμβάνει και ένα γενικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχε λεχθεί στην πρόταση του 2012 για, το, στο διάστημα 2012-2015 για την ευσορία των ζώων, που ήταν απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής. Επίσης, τίθεται ένα ακόμα ζήτημα το οποίο θέλω να αναφέρω. Πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Γεωργίας. Στα πλαίσια της, κοινής, της μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει, η προστασία των ζώων. Γιατί η προστασία των ζώων είναι απαραίτητη και για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων αξιών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε μια γενικά αηφόρο ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πρότυπα τα οποία θα είναι υψηλού επίπεδου για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε αυτό, σημαίνει ότι και τα προϊόντα μας θα μπορούν να ανταγωνίζονται με επωφελή τρόπο στις παγκόσμιες αγορές τα προϊόντα άλλων χωρών. Και αυτό αναφέρεται και στην εκθέσή μας. Θέλουμε τα πρότυπα αυτά τα οποία έχουμε θεσπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν σιγά σιγά παγκόσμια στάνταρτ, αλλά υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν επιτρέπουν προς το παρόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό σημαίνει ότι ορισμένα προϊόντα τα οποία εισάγουμε από τρίτες χώρες θα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια προβληματική που την έχουμε αναφέρει σε διάφορα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έχουμε αναφερθεί στον τρόπο ε, εκτροφής των ζώων στα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ε, διαδικασίες εκτροφής και επίσης για τα προβλήματα που συνάπτονται με την εισαγωγή ε, των προϊόντων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα οικιακά ζώα επίσης έχουμε θέσει μια σειρά από προτάσεις. Και επίσης, θέτε το ερώτημα των διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη χρήση φαρμακευτικών ε, σκευασμάτων στα ζώα, γιατί αυτό έχει και επίπτωση στα ανθρώπινα, ανθρώπινη υγεία και είναι πρότυπα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν. Και επίσης, άμα δούμε την ε, ε, διαδικασία παρα, παραγωγής τροφίμων υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην ευζοία των ζώων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση υπερβολικών αντιβιωτικών, ορμονών κτλ. Και επίση το θέμα της, των πειραμάτων τα οποία γίνονται στα ζώα και εκεί τίθεται το θέμα αν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να, προστατευτούν τα, ή, να προστατευτεί η ευζοία των ζώων. Όλα αυτά τα πειράματα θα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι λυσιτελής και να μην οδηγεί σε βάσανο των ζώων, γιατί η υγεία των ζώων είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο κύριε Ανδρουκάητη. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα ε, διαφέρει εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και συμμερίζω με την ανησυχία πολλών Ευρωπαίων για την σωστή μεταχείριση των ζώων. Η στρατηγική της Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς θέλουμε λοιπόν τώρα να ε, προβούμε στην ολοκλήρωση των αναπομενουσών ενεργειών. Αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη επιβολή των υφιστάμενων κανόνων, να βελτιώσουμε το διάλογο με του διαφόρου φορεί και να βρούμε τρόπου οι παράμετροι τη καλή διαβίωση των ζώων να ενταχθούν στι διεθνεί μα δραστηριότητε. Ό,τι αφορά την επιβολή τη νομοθεσία, η Ένωση διαθέτει μια δέσμη μέτρων και κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων που αφορούν πολλά, ε, πολλές κατηγορίες ζώων και πολλές δραστηριότητες, μεταφοράς φαγή, ε, δοκιμές σε ζώα κτλ. Αλλά και προϊόντα, ε, προϊόντα φώκιας, ζωοτροφές κτλ. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα στην πράξη και να διδαχθούμε από την εμπειρία των τελευταίων ετών. Άρα να εστιάσουμε στην καταπολέμηση της ε, μη συμμόρφωσης. Ε, θα προσπαθήσω να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση, να σταματήσουν ε, κάποιες πρακτικές σε ό,τι αφορά τους χείρους που τους κόβουν την ώρα και θα περιμένω και την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος για τις βέλτιστες πρακτικές μεταφοράς των ζώων που έχει στηριχθεί από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο το 2015 στο 2018 είναι ο χρονικός ορίζοντας αυτού του προγράμματος. Επίσης υπάρχει πρόταση της Κομισιόν για αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους επίσημους ελέγχους και έτσι θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή των προποθέσεων και απαιτήσεων για την καλή διαβίωση των ζώων. Παραδείγματο χάρη με τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Αναφορά για την καλή διαβίωση των ζώων. Σε ό,τι αφορά το διάλογο μεταξύ των αναφορέων, θα ήθελα να υπάρχει διάλογο μεταξύ ε, ενό ευρέω φάσματο ενδιαφερομένων φορέων. Θα κάνω μια πρώτη προσπάθεια για να δω κατά πόσον η κοινότητα φαίνεται να έχει όρεξη για μια τέτοια ε, άσκηση, για ένα τέτοιο εγχείρημα και μετά θα δούμε πώς μπορούμε αυτό το διάλογο να τον διαρθρώσουμε για το μέλλον. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διεθνή δράση, Υπάρχει ανησυχία ε, μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών για την ε, μεταχείριση των ζώων, αλλά δεν σταματά εντό των συνόρων μα αυτή η ανησυχία και πολύ σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να προωθούμε τη δική μα προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο για να προστατεύσουμε και την ανταγωνιστικότητα ε, τη κτηνοτροφία μα, που έχει καταβάλει τόσε πολλέ προσπάθειε τα πρόσφατα χρόνια για αυτά τα ζητήματα. Με τι προσπάθειε αυτέ μπορούμε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο τα ευρωπαϊκά πρότυπα παρά τι πιέσει τη παγκοσμιοποίηση μαζί με τους συναδέλφους μου που είναι αρμόδιοι για τη γεωργία και το εμπόριο εξετάζω τρόπους ε, για την ε, καλύτερη αξιοποίηση όλων των διατάξεων περί καλής διαφύσης των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε ένας παγκόσμιος ηγέτης ε, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη θέση μας για να ε, εκμεταλλευτούμε και καλύτερα τις αγορές που απαιτούν μια ε, σωστή δεοντολογία και ηθική παραγωγή και κτηνοτροφία. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει εντός του 2016 ε, μια νέα έρευνα ευρωβαρόμετρου για την καλή διαβίωση των ζώων που θα αποτελεί μια πολύ χρήσιμη πηγή πληροφοριών, ιδίω στους τομείς της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της εκπαίδευσης, κατάρτισης. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε τα επόμενα βήματα και βέβαια αφού θα έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου τα οποία θα αναλύσουμε και θα σας ενημερώσουμε γι' αυτά. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ Επίτροπε. Ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Ντες. Δεν είναι μέσα στην αίθουσα όμως. Οπότε θα περάσω στον επόμενο ομιλητή για ένα λεπτά, ο κύριος Δεκάστρο. Πρόεδρε, η Επιτροπή Γεωργίας έχει εκφράσει την ευαισθησία της σχετικά με την ευημερία των ζώων. Το επίπεδο προστασίας της ευημερίας αυτής είναι το υψηλότερο στον κόσμο. Η στρατηγική 12-15 ολοκληρώνεται και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τις προθέσεις της για την πιθανή νέα στρατηγική της. Πριν ζητήσουμε την ύπαρξη νέων κανόνων θα θέλαμε να μάθουμε ποιες είναι οι δράσεις της παρούσης στρατηγικής που δεν εφαρμόστηκαν ακόμα και αν υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει για την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή της. Να προσθέσω εδώ ότι αυτή τη στιγμή ζητούμε κανόνες όλο ένα πιο δεσμευτικούς για τους ε, κτηνοτρόφους μας, χωρίς να τεθεί το θέμα της αμοιβιότητας, τότε επιβαρύνουμε το παραγωγικό μας σύστημα και πολλές φορές κάποιες κτηνοτροφικές διαστηριότητες τις διώχνουμε από την Ευρώπη κατεβάζοντας το επίπεδο ευημερίας των συγκεκριμένων ζώων. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό James Nicholson. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η πολιτική μας για την ευζοία των ζώων θα πρέπει να ακολουθεί τις επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες και θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσει την πρακτική ανάγκη της παραγωγής τροφίμων. Και όχι βέβαια από την κοινή γνώμη και από ιδεαλισμό. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε την καλύτερη λύση για τα ζώα είναι να έχουμε μια λογική και εφαρμόσιμη στρατηγική η οποία να μην οδηγεί σε ιδιαίτερο αχθός για τους παραγωγούς. Πρέπει να καταλάβουμε τις συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν για τους παραγωγούς και τις ε, αθέλτες συνέπειες οι οποίες μπορούν να προκύψουν από ορισμένα μέτρα. Παραδείγματο χάρη, η Κομισιόν προτείνει, <clears throat> κάνει προτάσεις για τα, τη χρήση φαρμακευτικών συσκευασμάτων, αλλά αυτό θα μπορούσε να, έχει, να οδηγήσει σε προβλήματα στην υγεία των ζώων, <clears throat> εάν μειωθεί η χρήση φαρμακών. Επίσης, θα πρέπει να αναγνωριστεί και η σημασία της ε, προτίμησης των καταναλωτών. Στην ε, δική μου περιοχή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ορισμένα προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές έχουν ζητήσει να απαγορευτούν για να μπορέσει να υπάρξει προστασία των ε, προτύπων προστασία των ζώων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στις ε, εμπορικές μας συμφωνίες με άλλε χώρε. Δεν μπορούν οι χώρες, οι τρίτες χώρες να έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί δεν υπόκειται στα ίδια πρότυπα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διάφορε ασθένειε που πλήττουν τα βόηδη είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε μεγάλη πίεση στους ε, γεωργούς και εδώ κυρία Πρόεδρε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι μόνο τι γενικέ ρήτρε, αλλά και τον τρόπο εφαρμογή του. Ο κ. Φέντελ για μισή λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί βλέπω η πρόταση αυτή έχει προχωρήσει και έφτασε στην παρούσα φάση. Ε, κάποιες από τις προτάσεις της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων είναι δικές μας και περιλαμβάνονται, επαναλαμβάνω, στο κείμενο, στην πρόταση της Επιτροπής. Θα θέλαμε ε, επίσης ε, να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη προφορική ερώτηση και από ένα ψήφισμα και μια πλήρη συζήτηση. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ανδρουκάητης υπογράμμισε τους τομείς τους οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε σε λήψη μέτρων. Απαιτείται μια σαφέστατη αξιολόγηση αυτού τα οποία είχαμε, αυτών τα οποία είχαμε εντάξει στην προηγούμενη στρατηγική. Έτσι μόνο θα αναγνωρίσουμε τις πραγματικές μελλοντικές ανάγκες. Όπως είπε ο κύριος Νίκολσον, απαιτείται ένα ενιαίο πακέτο, καλά ισορροπημένο. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους ε, Ευρωπαίους Γεωργούς. Θα πρέπει να μην πάρουμε μέτρα εις βάρος των Ευρωπαίων Γεωργών, αλλά μαζί με αυτούς. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια ευρύτερη, θα έλεγα, ένα ευρύτερο πεδίο, μια ευρύτερη προοπτική και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σωστά έτσι ώστε να εναρμονίσουμε τις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς. Ε, ε, έχουμε μια ενοποιημένη εν πωλής αγορά, αλλά έχουμε και εντελώς διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις και ξέρουμε ότι οι οδηγίες δεν εφαρμόζονται όλες με τον ίδιο τρόπο. Στην ε, Σουηδία υπάρχει μια νομική ρύθμιση η οποία καλύπτει την παραγωγή χείρων που θα ίσχυε μέχρι το 2013. Αν δει τις μελέτες που έχουν γίνει στα πανεπιστήμια που ασχολούνται με την γεωργική παραγωγή, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Μόνο λίγες χώρες την έχουν εφαρμόσει. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις αντιβιωτικές ουσίες και πώς αυτό επηρεάζει τον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης ε, του κρέατος των ζώων αυτών. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει χώρος ο οποίος θα πρέπει να ερευνηθεί ακόμα και πρέπει να παρασκευαστούμε σωστότερα. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό κυρία Χάζερκαμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς επιβάλλουμε τεράστιο πόνο στα ζώα και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Υπάρχει και η βάση στο άρθρο 13 της συνθήκης που προβλέπει ότι τα ζώα είναι όντα συνειδητά και θα πρέπει να την χάνουν του απαιτούμενου σεβασμού. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καλύπτουν τις ανησυχίες μας αυτές. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη ουσιαστικά προστατεύει τις ταυρομαχίες ή και ε, ακόμα και άλλες απαράδεκτες αποκρουστικές πρακτικές. Συνεπώς λοιπόν ε, θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε και να αντιμετωπίζουμε έτσι τα ζώα, δεν θα πρέπει να τα με τέτοιο τρόπο ε, μέσα σε ε, φορτηγά, θα πρέπει να, στα, να σταματήσουμε την παραγωγή φουαγκρά με τον τρόπο τουλάχιστον που το κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φοβάμαι δεν προτείνει μια νέα στρατηγική και μάλιστα το είπε και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις πριν γίνει κάνει συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει ότι σέβεται το Κοινοβούλιο και σέβεται τις αρχές μας γύρω από την προστασία των ζώων. Um, Ευχαριστώ. Μόλις ήρθε ο κύριος Ντες στην αίθουσα. Θα του δώσω για δύο λεπτά το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα. Περίμενα δύο μοναχά ώρες για να μπορέσω να περάσω στα σύνορα. Εξ ονόματος του ΕΛΚ εγώ δίνω εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι η Κομισιόν έχει αναπτύξει μια νέα στρατηγική για την ευζοία των ζώων το επόμενο χρονικό διάστημα 2016-2020. Εμεί ω Γεωργοί γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ευζοία των ζώων που έχει μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα για μα. Μόνο τα ζώα τα οποία ανατρέφονται σωστά και έχουν σωστή υγεία θα φτάσουν υγιεί και στο πιάτο. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τον ρόλο της ευζοίας των ζώων στην γεωργία και να αναπτύξουμε τις σωστές στρατηγικές προστασίες. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένες αμφιβολίες. Δεν πρέπει τα μέτρα αυτά να οδηγήσουν στο ότι η παραγωγή της Ευρώπης να είναι λιγότερο ανταγωνιστική με τις παραγωγές άλλων χωρών. Η αύξηση της παραγωγής κρέατος στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 6% σε άλλες χώρες, ιδίω σε ασιατικές χώρες, έχει αυξηθεί κατά 300%. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να παραλείψουμε να προστατεύσουμε και την ευρωπαϊκή γεωργία και εκτινοτροφία. Προφανώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευζοία των ζώων, αλλά δεν πρέπει να καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή και ιδίως τις μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι ακριβώς αυτές οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να προστατευτούν. Ένα παράδειγμα. Όταν υπήρξαν ε, απαγορεύσεις σε σχέση με το κρέας, με το βόλιο κρέας λόγω της ε, ε, λόγω επιζώτιων, τότε ήταν πάρα πολύ μικρέ τέτοιε μικρέ επιχειρήσει οι οποίε αναγκάστηκαν να, να κλείσουν. Ένα λεπτό, κύριο Στέιλορ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό για την ε, ευζοία των ζώων από την διαπαραταξιακή ομάδα για τα ζώα, τη οποία είμαι πρόεδρο, είναι ένα ψήφισμα το οποίο στοχεύει ακριβώ στα κύρια θέματα που μα ενδιαφέρει. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι <clears throat> να έχουμε μια στρατηγική η οποία θα είναι υποφελής. εννέα μονάχα από τις 19 προτάσεις της Κομισιόν για δράση έχουν εφαρμοστεί. Γι' αυτό οποιαδήποτε νέα στρατηγική θα πρέπει με τρόπο στεναρό και κατεπήγοντα να ζητά να υπάρχει μια ε, νομοθεσία πλαισίου για την ευσοία των ζώων η οποία βελτιώνει τα πρότυπα στον τομέα αυτό και δεν τα αποδυναμώνει <clears throat> τα προηγούμενα μέτρα. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι όταν μιλούν ορισμένοι για την απλοποίηση των κανόνων, αυτό το οποίο κατά βάση εννοούν είναι η αποδυνάμωση των κανόνων. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι καλύτερη εφαρμογή. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στην πρόταση αυτή ψηφίσματος ώστε να μπορέσω να τα διεξέλθω όλα. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη να καταλάβουμε ότι τα ζώα είναι συνειδητά όντα και ότι τα ζώα υποφέρουν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά τα πρότυπα για την υγεία των ζώων ακολουθώντας τα ανθρώπινα πρότυπα. Και τέλος, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή εφαρμογή των κανονισμών. Η ευζοία των ζώων είναι ένα από τα τρία πιο προεξάρχοντα θέματα για τα οποία λαμβάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην περιοχή μου. Οι πολίτε μα νοιάζονται για τα ζώα και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα προστατεύσει. Ο κ. Άγνιου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Μιλάμε για καλή διαβίωση για ευζοία των ζώων. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Ε, Παραδείγματο χάρη, στην Νότια Ευρώπη διασκεδάζουν πολύ με τις σταυρομαχίες. Θα μπορούσε κανείς να πει ε, αν είσαι στη Ρώμη κάτω όπως οι Ρωμαίοι. Δυστυχώς όμως ε, έτσι λειτουργεί η ΚΑΠΑ. Οι Βρετανοί φορολογούμενοι επιδοτούν αυτές τις δραστηριότητες ε, γιατί επιληρώνουν για αυτές τις δραστηριότητες και σίγουρα περιλαμβάνεται αυτό στην νομοθεσία και έχουν υπάρξει και τροποποιήσει. Αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που να λέει για του Ορτανού φορολογουμένου ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα χρήματά του ε, για αυτέ τι δραστηριότητε. Θα ήθελα όμω να σα προειδοποιήσω ότι έρχεται δημοψήφισμα στη Βρετανία πολύ σύντομα για τη συμμετοχή τη στην Ένωση και δεν υπάρχει τίποτα ε, που να τους ε, δημιουργήσει περισσότερα ρίγη στους ε, Βρετανούς άνακουν που πηγαίνουν τα χρήματά τους. Και σε ό,τι αφορά τη θανάτωση των ζώων είναι ένα θέμα. Οι σκύλοι ε, που θανατώνονται για παράδειγμα, μετά τι τους συμβαίνει, τους θάβουν. Γιατί αυτό με ανησυχεί πιο πολύ το τι θα γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για το κατά να αποτεφρώνονται ή θάβονται. Έχουμε και την ε, περίπτωση των αερίτου του θερμοκηπίου. Ε, μήπως τα σφάγιά τους ε, τα χρησιμοποιούν μετά ως άλευρα ή ως ελίπασμα ή μπαίνουν ως πρωτεΐνη στις ζωοτροφές. Ε, αυτοί οι σκύλοι που μπορούν να από την Ανατολική Ασία έχουν πάνω από 20% λύσα. Δεν σημαίνει ε, ότι δεν μπορεί να έρθει και στην Ευρώπη αυτή η αρρώστια μαζί με τους ε, ανθρώπους που έρχονται από εκεί εφόσον ανοιχτά τα σύνορα. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η στρατηγική για την ευημερία των ζώων 2012-2015 ολοκληρώνεται. Χαίρομαι που το θέμα αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη και ελπίζω να υπάρξει μια νέα στρατηγική 15-20. Το άρθρο 13 λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ευημερία των ζώων διότι είναι ε, όπως είπαμε ευαίσθητες, ε, υπάρχει ευαίσθητα όντα. Δυστυχώς όμως και στον χειρουργικό τομέα ο πολλαπλασιασμός των εντατικών κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα μετά από την υπογραφή του TTIP, θα απειλήσει πάρα πολύ τις ε, αρχές μας. Ε, ε, εγώ έχω καταδικάσει κάποια παραδείγματα όπως ε, των χιλίων βοηδών στην Αρντές ή των χιλίων διακοσίων επίσης βοηδών στην Αλσατία. Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι απαράδεκτες. Είναι απαραίτητο λοιπόν και με τα μέσα τα οποία παρέχει η επιστήμη και λόγω επίσης των λίγων αποτελεσμάτων των πειραμάτων εις βάρος των ζώων να απαγορευτούν τα πειράματα αυτά και να αντικατασταθούν από εναλλακτικέ μεθόδους. Υποφέρουν φρικτά τα ζώα τα οποία δεν εξουδετερώνονται και δεν ε, ε τους αφαιρείται η συνείδηση από, δεν, αποευαισθητοποιούνται. Ε, αυτό είναι απαράδεκτο θα πρέπει να καταστεί ε, υποχρεωτική η αποευαισθητοποίηση επίσης ε, ε, και στα ζώα τα οποία παίρνουν μέρος σε ταυρομαχίες όπως επίσης και στα ζώα τα οποία σφάζονται με τελετουργικό τρόπο. Θα πρέπει όσοι παραβιάζουν τις ρυθμίσεις αυτές να τιμωρούνται, να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις εις βάρος τους. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ακολουθούν τις βέλτιστες ε, πρακτικές για ε, την, ε, για την αντιμετώπιση των σκύλων που ζουν ελεύθεροι στις περιοχές μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω ιδιαίτερα αυτή την αίτηση για μια ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016-2020 όπως και οι άλλοι ομιλητές πριν από μένα θεωρώ ότι η ευζοία των ζώων είναι πάρα πολύ σημαντική <clears throat> πρέπει να είναι χωρίς σύνορα αυτή η ευζοία και αυτό απαιτεί εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά αυτό πρέπει να είναι και προς όφελος των παραγωγών. Στην Αυστρία, στη χώρα μου, εμείς έχουμε πάρα πολύ ε, υψηλά επίπεδα προστασίας για την ε, ε, προστασία των ζώων, παραγωγός για τις οοτόκες όρνηθες, αλλά επίσης και σε ό,τι αφορά την μεταφορά των ζώων, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα πρότυπα, αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τηρούν απόλυτα αυτές τις προδιαγραφές και ιδίως για τη μεταφορά των ζώων γνωρίζω ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα λόγω του ανταγωνισμού και όπως είπαν και άλλοι ομιλητές που ανέφεραν τα θέματα αυτά ότι εμείς δεν βοηθούμε την ε, προστασία των ζώων εάν επιτρέπουμε τέτοιες πρακτικές. Και αυτό επίσης θα πρέπει να ισχύει και στην εμπορική μας πολιτική έναντι των τρίτων χωρών. Θα πρέπει να εξετάζουμε κάτω από ποιες παράγονται τα προϊόντα αυτά τα οποία φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Και είναι φανερό ότι πολλές φορές τα προϊόντα αυτά παράγονται με πολύ χαμηλότερα πρότυπα <clears throat> προστασίας των ζώων και έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ χαμηλότερο κόστος δημιουργώντας ανταγωνισμό. Θέλω λοιπόν να κάνω μία έκκληση να έχουμε ακόμα περισσότερες προδιαγραφές για την προστασία των ζώων αλλά θα πρέπει επίσης να κάνουμε και τις απαραίτητες ενέργειες, να πληροφορήσουμε καλύτερα τους καταναλωτές και να εξηγήσουμε ότι η μεγαλύτερη προστασία σημαίνει και υψηλότερο κόστος και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνεκτική και συνεπή εφαρμογή των προδιαγραφών προς το συμφέρον των παραγωγών και των καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Ο κ. Κόφωτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά μιλάμε για την προστασία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνουμε όμως τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε τα ζώα μας <clears throat> να ε, εκτρέφονται με έναν τρόπο ο οποίος <clears throat> δεν είναι βασανιστικού χαρακτήρα και δεν πρέπει να δεχόμαστε να γίνεται αυτή η παραβίαση των προδιαγραφών στην Δανία το ε, χείρον την χάνουν αποκοπής τη ουράς τους. Και <clears throat> υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία κατά των χωρών που θα πρέπει να λειτουργήσει εναντίον χωρών που παραβιάζουν τα ανθρωπίνα τα δικαιώματα των χωρών και επίσης εναντίον των χωρών που εφαρμόζουν μεταφορές μεγάλων αποστάσεων για τα ζώα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέγει πρόεδρο. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της ημερήσιας διάταξης, ένας συνάδελφος είπε ότι εμείς έχουμε προβλήματα με τρομοκράτες στην Ευρώπη, οπότε το να μιλάμε για την ευημερία των ζώων Ε, νομίζω ότι δεν, δεν τίθεται το δίλημα να διαλέξουμε ανάμεσα στην τρομοκρατία ή την ευημερία των ζώων. Η ευημερία των ζώων είναι ανθρώπινη και ευρωπαϊκή αξία, τμήμα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας των ζώων στον κόσμο και νομίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης θέλει να συνεχιστεί η διαδικασία βελτίωσης του επίπεδου αυτού. Η πλειοψηφία αυτή κατανοεί το τι σημαίνει η προστασία των ζώων και η ευημερία των ζώων για την ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα. Η έλλειψη λοιπόν μιας νέας στρατηγικής για τα ζώα το 2015 με 2020 είναι ένα πάρα πολύ κακό μήνυμα ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να συνεχίσει την πολιτική που ακολούθησε μέχρι τώρα για την βελτίωση ε, των τρόπων αντιμετώπισης των ζώων. Συνεπώς λοιπόν γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική αυτή και να προετοιμάσει τη νέα στρατηγική. Ο Γκάντι είπε ότι η μεγαλοσύνη των εθνών κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζώα. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς με τη νέα στρατηγική μπορούμε να αποδείξουμε την ανθρωπιά μας και την ηθική μας. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Γιάκοβτσίτς πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν συζητούμε την πολιτική για την ευζοία των ζώων πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα ζώα έχουν αισθήματα νιώθουν πόνο. Έχουν παρόμοια αισθήματα με τον άνθρωπο. Και αυτή πρέπει να είναι η αφετηρία μας και σε αυτή τη συζήτηση. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε σε αυτά τα ζώα. Όταν τα εκτρέφουμε, όταν δυστυχώς τα κλωνοποιούμε και όταν τα μεταφέρουμε με, το σωστό ή με σωστό τρόπο από μια περιοχή στην άλλη. Έτσι πρέπει να κατανοήσουμε και να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τον τρόπο μεταφοράς και την κλωνοποίηση των ζώων. Φυσικά χρειάζεται μια νέα στρατηγική. Η νέα αυτή όμως στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε και τα άγρια ζώα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε άγρια ζώα στο παράνομο, μάλλον ε, στα τσίρκα ή τα διαθέτουμε παράνομα στο εμπόριο. Επίσης τα κατοικίδια, ε, σκυλιά, γατιά, συχνά υφίστανται κακοί, κακομεταχείριση, κακοποιούνται και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να μας αντιμετωπίσει, να μας απασχολήσει. Η ισχύουσα στρατηγική λίγη φέτος. Σίγουρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για την περίοδο μέχρι το 2020 περιμένουμε να έχουμε τη σχετική πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Κάιτλης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ευθύνη από τη συνθήκη της Λισαβόνας να λάβει υπόψη την ευζοία των ζώων. Αλλά τα ζώα αυτή τη στιγμή υποφέρουν από τη μαζική εκτροφή, από τον τρόπο μεταφορές, από τα πειράματα σε ζώα, από τον τρόπο θανάτωσής τους. Κάθε χρόνο σκοτώνουμε εκατομμύρια ζώα κάθε χρόνο και η έλεγχοι είναι ελάχιστη. Δεν κολλάζονται οι παραβιάσεις. Δεν υπάρχει και καμία ε, ρύθμιση για τη μαζική εκτροφή ε, κουνελιών. Πότε θα τα αλλάξει λοιπόν αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε θα μπορέσει να προχωρήσει. Η στρατηγική η οποία εκπνέει εφέτος δεν έχει φέρει αποτελέσματα ούτε τα μισά από αυτά τα οποία προ... προέτρεπε. Θα πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν την εκτροφή των ζώων σε κλοβούς. Θα πρέπει να σταματήσουμε τα τεστ σε ζώα όταν υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι. Και επίση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε εμπορικέ συμφωνίε θα γίνεται η τήρηση των δικών μα προτύπων για την εκτροφή των ζώων. Ζητώ από την Κομισιόν να αγωνιστεί για μια πραγματική στρατηγική για την ευζοή των ζώων. Δεν έχει νόημα, είναι απαράδεκτη μια καρστέση. Οι πολίτε τη Ευρώπη δεν πρόκειται να αποδεχτούν κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα I can't stand the pain anymore. Αυτή είναι η κατάσταση των ζώων σήμερα. Σταματήστε λοιπόν να γράφετε μονάχα ε, κανόνες και τέτοια. Πηγαίνετε να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα των ζώων. Είναι ένα ηθικό θέμα το οποίο εμπλέκει όλους τους πολίτες τη Ευρώπης. Ευχαριστώ. Κύριε Εκ, θα δεχτείτε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Ντες. Κύριε Ντες, 30 δευτερόλεπτα. Έχω ένα ερώτημα για σας κύριε, Ντε, κύριε Εκ. Εσείς θα πρέπει να ξέρετε ότι εκεί που εσείς οι πράσινοι είχατε την εξουσία στα κρατήρια της ε, Γερμανίας, εκεί ήταν οι μεγαλύτερες εντατικές εκτροφές ζώων. Ενώ <clears throat> στην Ανατολική Ευρώπη δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε ένα τέτοιο φαινόμενο, κύριε Εκ. Το κεφάλαιο πηγαίνει πάντα εκεί που είναι πιο εύκολες οι ευκαιρίες για κερδοφορία. Στην Ανατολική Γερμανία υπήρχαν ευκαιρίες μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού που δημιουργήθηκαν. Αλλά από πού ήρθαν οι επενδυτές στην Ανατολική Γερμανία, πάρα πολύ από την Ολλανδία. Και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη. Δεν έχει να κάνει με το κόμμα το οποίο έχει την εξουσία. Και αυτό δεν έχει καμία απολύτω σχέση με αυτά που λέμε σήμερα για την προστασία των ζώων, η κομματική τοποθέτηση. Για ένα λεπτό, κύριο Ντυρό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, η στρατηγική 2012-2015 λύγει και είναι ε, διφορούμενο ο απολογισμός, αμφίσιμος. Ε, δεν ξέρω τι μας προτείνει η Κομισιόν για την περίοδο 2016-2020, νέα μέτρα, νέες στρατηγικές, μιλάτε για μια δημοσκόπηση, για μια έρευνα, αλλά Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαπραγματεύεται την διατλαντική εταιρική σχέση και μιλάμε για την εντατική κτηνοτροφή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εμείς θα πρέπει να νομοθετήσουμε ή όχι αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει συγκέντρωση. Είναι κλεισμένα τα ζώα. Ζουν σε συνθήκες ε, δουλείας. Θα πρέπει να απαγορευτούν αυτές οι συνθήκες εχμαλωσίας, συγγνώμη, τα ζώα. Θα ε, διαρωτηθούν πολύ σωστά οι πολίτες μη υποστηρίζουμε τους μεγάλους ομίλους και δεν θέλουμε τελικά τόσο να προστατεύσουμε τα ζώα και την ανθρώπινη υγεία. One Κύριος Τσούλο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνθήκη στο άρθρο 13 και ακούστηκε ήδη αυτό, λέγει ότι το θέμα της ευημερίας των ζώων θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια αντιμετώπισης συνειδητών όντων. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε λοιπόν υποκριτές και θα πρέπει αυτά τα οποία αποφασίζουμε να τα σεβόμεθα. Είμαστε υποκριτές λοιπόν σε επιστημονικό επίπεδο όταν χιλιάδες ζώα υφίστανται βασανιστήρια για λόγους πειραματισμού δίθεν επιστημονικού. Επίσης είμαστε και για πολιτιστικούς λόγους ένοχοι διότι χρησιμοποιούμε τα ζώα στα τσίρκα. Είμαστε υποκριτές <clears throat> και για θρησκευτικούς λόγους όταν ακολουθούμε συστήματα σφαγής που δημιουργούν τρομερά προβλήματα και κάνουν τα ζώα να υποφέρουν χωρίς λόγο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι η νέα στρατηγική που είναι απαραίτητη θα πρέπει να έχει στο κέντρο ε, της ε, την ευημερία των ζώων ακριβώς σαν όντα συνειδητά. Για δύο λεπτά ο κύριος Μπούντα και ε, Επίτροπε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η υγεία, η δική μας, η υγεία των ανθρώπων εξαρτάται και από την υγεία των ζώων και η υγεία των ζώων εξαρτάται από την ευημερία των ζώων και από τον τρόπο με τον οποίο εκτρέφονται. Γι' αυτό λοιπόν οι προτάσεις τα τελευταία χρόνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σωστές και υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά οι προσπάθειες αυτές να ενισχυθούν περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να διασφαλίσει την επικοινωνία με τους καταναλωτές και με τους γεωργούς για να γνωρίζει τις ανάγκες τους και να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων πλευρών έτσι ώστε τα δικαιώματα όλων να γίνονται σεβαστά. Θα πρέπει λοιπόν να μην ασχολείται, να μην ε, λαμβάνει μόνο ε, μέτρα νομοθετικά, ε, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει μια σωστή και εκ του σύνεγγης παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών από πλευράς των κρατών μελών. Και εδώ φοβάμαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας στην ε, τροφιμική αλυσίδα εις βάρος των γεωργών και αυτό θα δημιουργήσει και στη μείωση των επενδύσεων περαιτέρω στον τομέα αυτό. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά προβλήματα και σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Στα πλαίσια του streamlining των νομοθετικών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να κάνουμε την ζωή των γεωργών δυσκολότερη και οι γεωργοί οι οποίοι ε, έχουν επιδείξει την υπευθυνότητα που απαιτείται θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζονται οικονομικά στα πλαίσια βέβαια της διεθνούς αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με ορθότερο τρόπο τις δυνατότητες ε, χρήσης πιστώσεων από πλευράς του κοινοτικού προϋπολογισμού, ιδιαίτερα για τη βελτίωση των επερσέ εξυγχρονισμένους και καινοτόμους τρόπους παραγωγής. Η κυρία Μίτση. Ευχαριστώ. Τα ζώα έχουν αισθήματα, νιώθουν, πονούν, υποφέρουν όπως και ο άνθρωπος. Δυσκολεύομαι να καταλάβω πόσο μπορεί κανείς ε, να μεταχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο ε, ανυπεράσπιστα όντα. Δυστυχώς όμως πολλοί πιστεύουν ότι τα ζώα ε, υπάρχουν απλά για να τα εκμεταλλευόμαστε, είτε για να τα τρώμε, είτε για να τα κυνηγούμε ή να τα χρησιμοποιούμε για την επιστήμη, είτε για άλλους λόγους. Δεν θα πρέπει όμως ε, να κακοποιούνται τα ζώα, θα πρέπει να τα σφερόμαστε με αξιοπρέπεια, δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν ε, για τη συμπεριφορά των ανθρώπων γιατί δεν έχουν φωνή. Εμείς πρέπει να τους δώσουμε φωνή. Και επειδή λύγει αυτή η στρατηγική το 2015, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να υλοποιήσει τα σημεία τη στρατηγικής αυτής που εκκρεμούν ακόμη και να καταρτήσει μια νέα στρατηγική προ όφελο των ζώων αλλά και όλων όσων ε, τα σέβονται και τα αγαπούν. Ας αποδείξουμε ότι είμαστε πολιτισμένοι και ας διδανίσουμε τη φωνή μας για να υπερασπιστούμε τα ζώα που χρειάζονται την προστασία μας. Ε, γιατί πολλές φορές ε, αγαπούν και συγχωρούν περισσότερο από ότι ο άνθρωπος. Κυρία Γκέρλινγκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερη επιβολή, συντονισμό των νομοθεσιών που ήδη υπάρχει είναι σημαντικό παράγοντα για να βελτιώσουμε την ζωή των ζώων. Σίγουρα ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, επιβιώσει η κτηνοτροφία, να στηριχθεί η παραγωγή ε, του κρέατος και να μην υπάρχει όμως η λεγόμενη διαρροή, δηλαδή περισσότερες εισαγωγές σε βάρος των δικών μας κτηνοτρόφων. Όλα αυτά θα προστατεύσουν και την καλή υγεία των ζώων. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, θα πρέπει η κακοποίηση να αποφευθεί, να βελτιωθούν οι κτηνοτροφικές συνθήκες, οι συνθήκες μεταφοράς, ε, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. μας είπε βέβαια και ο κ. Δέστη και την εμπειρία, αλλά πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και σε επίπεδο κρατών μελών. Εδώ πολλοί βουλευτέ είπαν ότι πολλά λέμε, αλλά λίγα κάνουμε για την καλή διαβίωση των ζώων. Δεν συμβαίνει όμω αυτό. Έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο. Α πάψουμε λοιπόν να, να μειώνουμε ε, του εαυτού μα. Απλά πρέπει να επιβάλλουν οι κυβερνήσει των κρατών μελών αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, κ. Στέρι Κάμπρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για να εξασφαλίσουμε μια πραγματική στρατηγική για την ευζοία των ζώων, θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η στρατηγική την βασική ιδέα η οποία διατρέχει την προστασία και την ευζοία των ζώων. Η ιδέα αυτή είναι μια φιλοσοφική και ηθική αξία που συνήθως δεν την αναφέρουμε. Συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ζώα γιατί έχουν δικαιώματα. και θα πρέπει να υπάρξει ίσως το σωστό συσχετισμός δικαιωμάτων και καθηκόντων. Θα πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα <clears throat> και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωρίζετε το δικαίωμά τους να έχουν δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα έγγραφά μας. Γιατί αυτή είναι η βάση επί τις οποίες εμείς οικοδομούμε την προστασία μας και τη στρατηγική για την ευζοία των ζώων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά η κυρία Σράιερ Πίλακ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αναφέρομαι στη συνέχιση της στρατηγικής για την ευημερία των ζώων. Εγώ είμαι κατά. Για ποιο λόγο. Οι οδηγίες και οι κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως. Τα μέσα επίσης που έχουμε μέχρι τώρα δεχθεί ε, και εφαρμόσει θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται πλήρως. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν έχει νόημα η Ευρώπη ε, να υιοθετούμε κανόνες εφόσον δεν εφαρμόζονται και δεν γίνονται σεβαστοί μόνο και μόνο για να αυξάνουμε το κόστος. Έχουμε συζητήσει θέματα όπως η γεωργική κρίση εδώ και νομίζω ότι αν τεθούν αυστηρότερες απαιτήσει από τους γεωργούς δεν οδηγούμεθα πουθενά. Μιλάμε για την ευμερία των ζώων ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για την ευμερία ευημερία των πολιτών μας. Αφήνουμε τους πρόσφυγες να ζουν μέσα στο κρύο και στο χιόνι και βάζουμε συστήματα θέρμανσης για τα ζώα και επίσης θέλουμε να περιορίσουμε και το όριο για τη μεταφορά ζώων από τις 8 ώρες στις 7. Αφήνουμε τον κόσμο να ζει στα χιόνια γιατί είναι άστεγος και ενώ τα ζώα πρέπει να έχουν φως, ζέστη και άλλα κομφόρ. Νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, Πρόεδρε, να αλλάξουμε ανατολισμό. Είναι η ώρα να στραφούμε στα πραγματικά προβλήματα, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Την κρίση του ασύλου, να βρούμε λύσεις για αυτήν και να αντιμετωπίσουμε επίσης τις επιθέσεις των τρομοκρατών και του ΝΤΑΕΣ. Νομίζω ότι τα θέματα θα πρέπει να είναι η προστασία των ανθρώπων. Έχετε δύο αιτήματα με μπλε κάρτες. Ε, ο ένας που ζητά να σας ερωτήσει έχει ήδη μιλήσει, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάρ. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στην κυρία Σράιδερ. Έχετε παρουσιάσει την εικόνα των γεωργών αλλά για μένα ε, νομίζω ότι είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύσει και τα οικιακά ζώα όπου δεν υπάρχει καμία ε, ε, κανένα συνεκτικό πλαίσιο και υποφέρουν τα ζώα και στα, στο οικιακό πλαίσιο. Τι πιστεύετε πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά. Χωρίς μικρόφωνο. Εσύ. Εγώ συμφωνώ ότι είναι σημαντικό το σημείο αυτό. Πολλές φορές έχουμε τονίσει στις ε, συστάσεις μας ότι πρέπει να ληφθεί και αυτό το στοιχείο υπόψη. Όλες <clears throat> οι πτυχές της προστασίας των ζώων θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτήν την ε, ε ρύθμιση. Η κυρία Κριστίνα Αγγιλέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι ολοκληρώνεται η δεύτερη στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων στα τέλη του έτους. Ε, έχουμε ε, τη δεύτερη αυτή στρατηγική και έχουμε πλέον ε, ένα οπλαστάσιο κανόνων που όμως δείχνει ότι έχουμε διαφορετική εφαρμογή. Έχουμε τους στόχους αυτής της στρατηγικής. Θα ήθελα να ξέρω όμως και τα αποτελέσματα. Χρειαζόταν να δούμε αυτά τα προβλήματα μήπως πιο ολοκληρωμένα με ένα κοινό πλαίσιο για την καλλιγεία των ζώων. Νομίζω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτή τη δεύτερη στρατηγική. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να ξέρω, όπω είπα, το αποτέλεσμα. Να δούμε πρώτα το αποτέλεσμα τη δεύτερη αυτή στρατηγική. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να δω είναι τι θα πει ε, ο Ευρωπαίος πολίτης ε, με αυτή την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για αυτά τα οποία συζητούμε εδώ και αν είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να πληρώσουν παραπάνω για την καλή υγεία των ε, ζώων και την καλή διαβίωσή τους. Επαναλαμβάνω, το βασικό με ενδιαφέρει είναι να δούμε το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι έχουμε πολλούς κανόνες, σωστούς κανόνες. Δεν ξέρω αν ε, ομοιόμορφα όμως ε, αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα τα κράτη-μέλη και θα δούμε και τις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Είμαστε ή δεν είμαστε τόσο απαιτητικοί και σε αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο κ. Κουσνίκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, να σας υπενθυμίσω ότι από τις 19 προτάσεις για μέτρα που είχε περιλάβει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο 9 μέχρι στιγμής έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Θα έπρεπε ίσως η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να καλύψει το χαμένο έδαφος και έχει νόημα να προτείνει νέα μέτρα πρέπει αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 να γίνουν πραγματικότητα. Και οι εκτροφείς ζώων στην Ευρώπη να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες <clears throat> και με τους ανταγωνιστές τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο και σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει επίσης στις συμφωνίες με τρίτα κράτη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει ότι θα λαμβάνεται υπόψη πλήρω η προστασία των ζώων. Υπάρχουν κανόνε που θα πρέπει να ισχύουν και για του εξαγωγείς ζωικών προϊόντων από τρίτε χώρε. Αλλιώ θα βρεθεί σε απειλή η δική μα παραγωγή. Ο κύριος Ντελέη. Η κυρία Ντελέη. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι τίθεται το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει πριν <clears throat> από τι προτάσει Ευρωπαϊκή είναι πολύ σημαντική η υγεία των ζώων. Οι πολίτες μας όλο και περισσότερο θέλουν να καταναλώνουν υπεύθυνα. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίσουν και την προέλευση αυτών των ζώων και τις συνθήκες κάτω από τις εκτρέφονται τα ζώα αυτά. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να χαιρετήσουμε τις προσπάθειε που έχουν γίνει σε διάφορου τομεί. Και φυσικά αυτό εμπλέκει και του. Ε, κτηνοτρόφους, <clears throat> οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν προς την παραγωγή ποιότητας. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεχίσει προσπάθειες για μια νέα στρατηγική για την ευζοία των ζώων, θα πρέπει να είναι αντικειμενική και πραγματιστική, να περιλαμβάνει το σύνολο των εμπλεκομένων, τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Δεν πρέπει να δακτυλοδεικτούμε μόνο τους παραγωγούς, αλλά να κάνουμε μια υποστήριξη των βελτίστων πρακτικών και να ενισχύουμε την πρόοδο. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μία πλευρά να ζητούμε την ευσοία των ζώων και από την άλλη μεριά να επιβάλλουμε δυσβάστακτο άχθος στους παραγωγούς. Θα πρέπει να είναι ρεαλιστική η νομοθεσία μας. Θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν το σωστό υπόδειγμα για την παραγωγή ζωικών προϊόντων στην Ευρώπη. Έχουμε εκθέσεις που δείχνουν το πόσο δύσκολο είναι να συνάπτονται οι βασικές ε, προθέσεις με τα αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Οι καταναλωτές θέλουν να έχουν και μείωση των αερίων θερμοκηπίου, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό με τον περιορισμό της εκπομπής μεθανίου από τις αγελάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντεμπαχ. Κυρία Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Παρά την κρίση που αντιμετωπίζουμε, η οικονομική κρίση, θα πρέπει να σκεφτούμε και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, ευζοίας των ζώων. Και το έχω τονίσει αυτό και προηγουμένως στα πλαίσια της εκπόνησης στρατηγικής 2012-2015. Τότε προσπάθησαν ορισμένοι να μας υποχρεώσουν να δεχτούμε κάτι λόγω της ε, οικονομικής κρίσης, το οποίο δεν συνάδει με την ευζοία των ζώων. Και σήμερα έρχονται άλλοι οι οποίοι μας λένε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις θα πρέπει να υπαγορεύουν τη στάση μας. Όχι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να δεχτεί κάτι τέτοιο. Παρά την κρίση, παρά την τρομοκρατία, όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Πρέπει να τηρηθεί το άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι είναι ε, ενσυνείδητα όντα τα ζώα και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποβάλει μια στρατηγική που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων αυτών. Γιατί όλα αυτά συνάπτονται φυσικά και με την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία των ζώων σημαίνει και υγεία των ανθρώπων. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα διαχωρίσουμε αυτά τα σημεία. Θα πρέπει να έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι Ευρώπη των ανθρώπων, αλλά αυτή η Ευρώπη πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα δικαιώματα των ζώων. Ο λόγος τώρα στον κύριο Ντάλτον. Ευχαριστώ. Έχουμε αυστηρότατους κανόνες για την ευημερία των ζώων, αλλά δεν έχουν καμία αξία εφόσον δεν εφαρμόζονται. Το θέμα είναι η εφαρμογή. Τι νόημα έχει μια νέα στρατηγική αν διαπιστώνουμε ότι δεν εξυπηρετούνται και δεν γίνονται αντικείμενο σεβασμού οι ισχύουσες ρυθμίσεις ε, σε κανόνες για τη μεταφορά των ζώων. Βλέπουμε ότι η πραγματικότητα απέχει από την νομοθεσία. Επίσης υπάρχουν προβλήματα και με παράνομες εισαγωγές. Μεταφέρονται ζώα των οποίων η υγεία είναι αμφισβητήσιμη. Συνεπώς λοιπόν δεν απαιτούνται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Νέες ρυθμίσεις που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε θα χειροτερεύσουν την κατάσταση. Θέλουμε η ισχύουσα νομοθεσία να εφαρμοστεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα του σεβασμού των ζώων. Τότε μόνο θα μπορέσουμε στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο να βρούμε λύσεις. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράγματι ιδιαίτερα ισχυρούς κανόνες. Η Ευρωπαίοι Γεωργοί νομίζω μπορεί να είναι υπερήφανοι για την κοινή αγροτική πολιτική τα τις τελευταίες δεκαετίες. Εγώ παρακολουθώ τα θέματα αυτά και στη Σλοβενία από κοντά. Είμαι Γεωργός και είμαι και τέος Υπουργός Γεωργίας Ξέρω τι περνούν, τι υφίστανται οι γεωργοί για να μπορέσουν να προσαρμοστούν ε, στις ρυθμίσεις οι οποίες απαιτείται να εφαρμοστούν στις ε, παραγωγές τους. Ε, επίσης υπάρχουν ειδικότερε απαιτήσει πολύ ισχυρές στον τομέα της παραγωγής χείριου κρέατος όπως επίσης και για την παραγωγή πουλερικών στην πτηνοτροφία. Πρέπει λοιπόν οι εγγυήσει τις οποίες θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οδηγήσουν σε ενιαίους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από με τους γεωργούς αλλά και με τους καταναλωτές. Μόνο έτσι θα κάνουμε βήματα με σωστό τρόπο. Δεν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως ε, ε, βιαστικοί θα πρέπει να δούμε ε, τι συμβαίνει επίσης και στις χώρες από τις οποίες εισάγουμε προϊόντα κρέατος. Νομίζω ότι αν ε, αφήσουμε ανεξέλεγκτες τις εισαγωγές, τότε θα θέσουμε τους Ευρωπαίους ε, κτηνοτρόφους σε εξαιρετικά κακή κατάσταση. Και νομίζω ότι οι πρώτοι που θα την πληρώσουν θα είναι οι μικροί κτηνοτρόφοι. Βλέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην παραγωγή ε, κρέατος προς Ρώση και στις ε, ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες εισάγουμε. Μπράνεν. Um, Ευχαριστώ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στρέφονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει αποφασιστική δράση για τη διατήρηση της ε, καλής διαβίωσης των ζώων που θα πρέπει να έχει ως αφετηρία αυτή τη νέα στρατηγική με ένα ε, σχέδιο για την καλή διαβίωση με μια μοναπευθυντική θηρίδα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή διαβίωση των ζώων. Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της ευζοίας των ζώων με συντονισμένο καλό τρόπο είναι, έχουν ε, ε, συνέστηση τα, τα ζώα, έχουν συνείδηση. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, έτσι ακούσαμε σήμερα. Και μόνο αν αντιληφθούμε τη βασική αυτή αλήθεια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο εντός Ένωσης αλλά και πέραν αυτής για να βελτιώσουμε την ε, καλή διαβίωση, να πάψουν εξαρτήσεις τρίτες χώρες ε, και να ε, καμφθεί το παράνομο εμπόριο εξωτικών κατοικιδίων και άλλων. Είναι πλέον καιρός να υιοθετήσουμε μια άλλη, μια νέα στρατηγική, πιο στεναρή. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι η κυρία Νόιχελ. Τίθεται το ερώτημα κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, γιατί δεν υπάρχει καμία νέα στρατηγική για την προστασία των ζώων. Ποιο είναι το, το υπόβαθρο αυτής της απουσίας. Όχι μόνο για την δική μας Επιτροπή που είναι αρμόδια για την προστασία των ζώων, αλλά και άλλες επιτροπές ξέρουν ότι δεν έχει γίνει αρκετή πρόοδο στα θέματα αυτά. Παραδείγματο χάρη το ίδιο συμβαίνει και για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Κομισιόν λοιπόν αρνείται, γιατί δεν δέχεται να θεσπίσει σαφείς στόχους, να ακολουθήσει ένα σαφή δρόμο, να ακολουθήσει ένα οδικό χάρτη που να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα για να υπάρξει πρόοδος στην Ευρώπη. Εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν αναφέρει οι συνάδελφοί μου εδώ είναι θέματα τα οποία η Κομισιόν τα παραγνωρίζει και δεν δίνει καμία σημασία. Χρειαζόμαστε ένα σαφές πλαίσιο, μια σαφή στρατηγική. Και εγώ δίνω μεγάλη σημασία στα θέματα της ε, κτηνιατρικής και θέλω να δίνεται ίδια σημασία στην κτηνιατρική όπως και στην ανθρώπινη ιατρική. γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σαφήνεια και μια στρατηγική. Ακολουθεί ο κύριος Σιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στον τομέα της ευημερίας των ζώων είναι σημαντικά και θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα σαφέστερο ίσως νομικό πλαίσιο γύρω από αυτά και να διασφαλίσουμε την συνοχή ανάμεσα, την συνεκτικότητα μάλλον των τρόπων χρηματοδότησης των μέτρων αυτών. Όπως ε, είπαν και άλλοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων στην Ευρώπη, κάτι το οποίο μερικές φορές είναι δύσκολο να ε, εφαρμοστεί. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο τι συμβαίνει στις τρίτες χώρες. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα οικόσιτα ζώα είναι απαραίτητο να καλυφθεί και η αυτή η κατηγορία. Ε, δεν υπάρχει ιδιαίτερα, ιδιαίτερη συνοχή θα έλεγα. στους τρόπους και στις ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο τομέα. Τζουφριντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η στρατηγική 2012-2015 επέδρασε θετικά και οι δράσεις που ανελήφθησαν για την βελτίωση της ευημερία των ζώων ήταν σαφείς. Ε, νομίζω ότι αυτό δείχνει την ευαισθησία που υπάρχει και ενισχύεται μάλιστα για την ευημερία των ζώων. Η κοινή γνώμη είναι πολύ πιο προοδευτική από τα ευρωπαϊκά όργανα και δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε τη συνέχιση συστηματικής βίασης βάρος των ζώων. Έχουμε στα πλαίσια του κανονισμού για την υγεία επίσης των ζώων ε, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικότατο για ε, τους, ε, και για τους ανθρώπους. Έχουν γίνει λοιπόν τα πρώτα βήματα και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Να διαμορφώσει μια στρατηγική η οποία να αντιμετωπίζει τις μορφές άσκησης βίας εις βάρος των ζώων. Ευχαριστώ. Πριν τη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ, ομιλητής, ο κύριος Σεράου Σάντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε για να εξασφαλίσουμε την υγεία των ζώων. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του να βελτιώσουμε την υγεία, τη σωματική και ψυχολογική υγεία των ζώων και να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των παραγωγών. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κανένα από τα δύο άκρα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ε, ευζοία των ζώων και επίσης και των ηχθείων. Σε περίπτωση ηχθειοκαλλιέργειας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες. Η Κομισιό λοιπόν θα πρέπει να μας δίνει στοιχεία για την επιστημονική έρευνα που έχει προκύψει από τη στρατηγική 2012-2015. Υπάρχουν και πορίσματα σε σχέση με την επίπτωση της αλίας στην ευζοία των νυχτιών. Θα πρέπει και όλα αυτά να ληφθούν υπόψη για το μέλλον. Ευχαριστώ. Υπάρχουν έξι βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο με την διαδικασία Catch the Πρώτος είναι ο κύριος Μυροσλάβου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούμε το θέμα της ευζοίας των ζώων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να το δούμε. Είτε μιλάμε για ζώα που εκτρέβονται σε συνθήκες εντατικής εκτροφής και τα οποία επομένως Ζούνε κάτω από συνθήκες πολύ ανθυγινές, αλλά και για τα οικόσιτα ζώα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Θα πρέπει και αυτά να ζουν σε καλές συνθήκες. Θα ήθελα επίσης να σκεφτούμε και τις μεθόδους φώνευσης των ζώων. και επίσης για τα θέματα δοκιμασιών και πειραμάτων που γίνονται στα ζώα. <clears throat> Πρέπει και εκεί να αποφεύγουμε να κάνουμε τέτοιες ε, ενέργειες. Και επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τη μεταφορά σε μεγάλη απόσταση των ζώων και επίσης και τα κλωνοποιημένα ζώα υποφέρουν φρικτά. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη στο Κοινοβούλιο. Να σας πενθυμίσω ότι η διαδικασία Catch the Eye είναι ομιλίες ενός λεπτού. Ο κύριος Καπούτο Νικόλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το υψηλό επίπεδο ευημερίας ή ευζοίας των ζώων είναι κάτι το οποίο θα δώσει εγγυήσεις και για την υγεία τους και θα βελτιώσει και την παραγωγικότητα της εκτροφής τους. Ε, η στρατηγική 12-15 επέτρεψε να γίνουν βήματα προς τα εμπρός, θα πρέπει όμως να υπάρξει μια πιο φιλόδοξη πολιτική για την προστασία περίοδο 16-20 με ένα απλοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι περίπλοκο το θέμα της ευζοίας των ζώων και υπάρχει και μία νομική αβεβαιότητα που δεν θα πρέπει να λειτουργεί αρνητικά για τους παραγωγούς. Ταυτόχρονα η ευκταία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιτρέψει την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που σέβονται τις ορθές πρακτικές ε, των κτηνοτροφικών τους μονάδων. Και θα πρέπει να καλύψουμε επίσης ε, και τα αδέσποτα ζώα ε, και τα οικόσιτα ζώα έτσι ώστε να πετύχουμε μια βελτίωση των όρων ζωής των συγκεκριμένων αυτών όντων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προστασία της ευζοίας των ζώων είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα που πρέπει να λάβει υπόψη της η επιτροπή. η στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2012 χιλιάδες έφερε αρκετά θετικά αποτελέσματα βοηθώντας στην εξάλληψη του φαινομένου βασανισμού των ζώων. συχνά όμως σε ολόκληρη την επικράτεια της ευρώπης συναντάμε βασανισμούς και κακομεταχείριση των ζώων. θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα ζώα κυριολεκτικά βασανίζονται και υποκύπτουν σε φρικτούς πόνους στο βωμό της εσχροκέρδειας όπως συμβαίνει με την φαλαινοθυρία. θα πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή επιτροπή να λάβει πολλαπλά πρόσθετα μέτρα με γνώμονα την καλή μεταχείριση των ζώων και φυσικά την προστασία αυτών από κάθε είδους πρακτικές βασανιστήριων ή ανάλογων πρακτικών που οδηγούν στην κακή μεταχείριση των ζώων. τέλος θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση για ένα απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων. ευχαριστώ. Thanks. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μίλλερ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ε, υποστηρίζω όλα αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι σε σχέση με την προστασία των ζώων. Αυτό πρέπει να είναι μια <clears throat> μεγάλη προτεραιότητα για όλους τους κατεκρινοτρόφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 30 χρόνια φυσικά έχει αλλάξει πολύ έντονα η διαδικασία εκτροφής των ζώων έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος αλλά υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη χρήση επενδύσεων για να υπάρξει εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των παχνιών των ζώων. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ε, στάση ε, και είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη πιστοποίηση των εγκαταστάσεων εκτροφής των ζώων. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτείται και χρειαζόμαστε να υπάρχουν και διαδικασίες εφικτές και απτές οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει όμως να απολέσουμε τις αγορές μας και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε είναι ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταχείριση των ζώων στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό χρειάζεται μια εναρμόνιση και να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο σήμα το οποίο δείχνει ότι τα ζώα έχουν εκτραφεί κάτω από καλέ συνθήκε, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ο κύριο Βιέγκος. Οι παραβιάσει τη ευζοία των ζώων είναι τα αποτελέσματα μια γεωργία η οποία όλο και περισσότερο υπόκειται στην λογική τη κερδοφορία μια παγκόσμια αγορά που γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστική η εντατικότητα της παραγωγής σε ό,τι αφορά παραγωγικά χάρη της, ε, τα κουνέλια ή τα γουρούνια ή τις κότες είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε βάσανα των ζώων και αυτό είναι αποτέλεσμα της ε, οικονομικής λογικής που υποχρεώνει τους γεωργούς να καταφεύγουν σε τέτοια εντατική γεωργία, εκτινοτροφία μάλλον, αλλιώς θα χάσουν τη δυνατότητα επιβίωσής τους. Όλα αυτά είναι αποτελέσμα μιας νεοφιλελεύθερης εκτινοτροφίας ε, που οθείται από τις αγορές και όπου το κέρδος είναι πολύ πιο σημαντικό από την ευζοία των ζώων και όλα τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία μας ε, έρχονται δείχνουν ότι έχουμε περάσει σε μια απόλυτη παραφροσύνη. Καταστρέφουμε την υγεία των ζώων, τη βιοπικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε την κτηνοτροφία μας σε μια άλλη κατεύθυνση που να σέβεται το, τη την ευζοία των ζώων και την ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Uh, η επικουρικότητα λέγει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται όσο συντομότερα γίνεται ε, στους πολίτες. Οπότε πάρα πολλά από τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα θα μπορούσαν να αποφασιστούν από τα ίδια τα κράτη-έθνη. Νομίζω ότι αυτή η γενική νομοθετική κανόνες δεν είναι απαραίτητη. Τα κράτη-μέλη να έχουν την δυνατότητα να τερματίσουν την εισαγωγή ζώντων ή νεκρών ζώων ε, στις ε, επικράτειές τους. Το ίδιο ισχύει και για τα λεγόμενα εξωτικά οικόσιτα και επίσης και τα λεγόμενα διακοσμη, τους λεγόμενους διακοσμητικούς ηχθείες. Είναι θέματα τα οποία επηρεάζουν ιδιαιτέρως ε, την οικονομική δραστηριότητα στη δική μου ε, εκλογική περιφέρεια. Νομίζω ε, ότι θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουμε το κρέας όπως αντιμετωπίζουμε τον καπνό και ότι ε, είναι κάτι το ανθυγινό γιατί έτσι προσβάλλει ε, τους κτηνοτρόφους με απαράδεκτο τρόπο. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Επίτροπο κύριο Αντρουκάητης. Έχετε το λόγο κύριε Αντρουκάητης. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Άκουσα πολύ προσεκτικά Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι δραστήρια στο θέμα αυτό της ευημερίας των ζώων. Άκουσα πάρα πολλές προτάσεις ε, για την ευζοία, άκουσα πολλές προτάσεις για τη νέα στρατηγική και επίσης για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ευημερία των Ζώων Όλες αυτές οι επιλογές αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές και βρίσκονται υποσυζήτηση από τις υπηρεσίες μου και το γραφείο μου. Και θα ξεκινήσουμε επίσης λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα οποία ε, στοιχεία μας δίνει το Ευρωβαρόμετρο. Το θέμα είναι να προσθέσουμε αξία στην τροφομική αλυσίδα σεβόμενη τα συμφέροντα των ε, εμπλεκομένων. Απαιτούνται νέες πληροφορίες οι οποίες θα γίνουν διαθέσιμες το 2016 και έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις θεμητές προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Η σωστή εφαρμογή επίσης του κοινοτικού κεκτημένου είναι μια βασική κομβική θα έλεγα προτεραιότητα και θα περιμένουμε την επόμενη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου και θα δούμε τα αποτελέσματα τα οποία μας δίδει ε, και τι ε, ρόλο μπορεί να παίξει στον συγκεκριμένο τομέα η σωστή πληροφόρηση των πολιτών. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυθμίσεων θα δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς για την ευζοία προωθώντας ε, τα συμφέροντα των εμπλεκομένων και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε στην ακτινοτροφία και να μπορέσουμε να βρούμε επίσης και νέες αγορές με υψηλά επίπεδα και απαιτήσει. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει ένα ψήφισμα από πλευρά σας σε εύθετο χρόνο και να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνει πολύ σοβαρά τα θέματα της ευημερίας των ζώων Αυτά τα θέματα ε, θα ανταλάβουμε υπόψη μας ε, και στο ε, άμεσο μέλλον για να προστατεύσουμε <coughs> την τροφιμική αλυσίδα πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε. Θα κατατεθούν προτάσεις ψηφίσματος για την ολοκλήρωση της συζήτησης αυτή.